Από την παράγραφο 8. Κατέθεσα τροπολογία διαγραφής για διάφορα στοιχεία, τα αναφέρω εντάχει. Όταν λέμε ότι ε, αυτές οι παράνομες εμπορικές ε, και καταχρηστικές ε, πρακτικές παρακολουθούνται επαρκώς. Θεωρώ ότι από την άλλη είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένες ε, χώρε ή ορισμένα ε, μέσα και αναφέρομαι εδώ στο, στο τι συνέβη με το EU Libor και το Libor. Μετά, στη 13. Είναι ένα στοιχείο επί εδώ. Νομίζω ότι η προστασία των καταναλωτών περνά από την ενσωμάτωσή του στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτή η υπόθεση, δηλαδή το 20% των το, διοικητικών συμβουλίων αποτελείται από καταναλωτέ, δεν ε, θεωρώ θετικό να υπάρξει ε, αυτός ο μηχανισμός. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό σε περίπτωση των εργαζομένων που συνεργάζονται μαζί με, τους, ε, με τις επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει όμως και με τους καταναλωτές. Μετά για τις υπόλοιπες τροπολογίες ε, προτείνω τη διαγραφή ε, στην παράγραφο 15 για τον μηχανισμό προσφυγής ε, μέσω εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Όχι επειδή διαφωνώ γενικά με την αρχή, αλλά επειδή δεν θεωρώ ότι συνάδει η διατύπωση με τα όσα ψηφίστηκαν στην Επιτροπή μας. Όμως ε, είδα ότι υπάρχουν 8 τροπολογίες που ε, έχουν κατατεθεί από συναδέλφους για αυτό το κομμάτι του κειμένου και όπως είπε ο εισηγητής σίγουρα θα βρούμε μια, μια ενδιαφέρουσα συμβαστική πρόταση. Επίσης, κάποια σημεία τώρα που είναι σημαντικά. Εδώ δεν μιλάμε για ε, διαγραφές πλέον, αλλά για προσθήκες που προτείνουμε με κάποιους συναδέλφους από το ΕΛΚ προτείνουμε ε, τροποποιήσεις ό,τι αφορά την πληροφόρηση που δίνεται στους καταναλωτές, ιδιαίτερα στο σημείο 4. Και πρέπει πράγματι να δούμε ε, αυτή η πληροφόρηση να είναι στοχευμένη και αν είναι αυτό δυνατό συγκρίσιμη και να μην πέφτουμε στην παραγίδα να έχουμε συνεχώς περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα δεδομένα, εφόσον ξέρουμε ότι από κάποια στιγμή και μετά ο καταναλωτής πλέον δεν μπορεί να χειριστεί όλες αυτές τις πληροφορίες. Πρέπει να γίνεται λοιπόν μια σωστή σύνθεση. Σημαντικό αυτό το στοιχείο. Σε πολλές φορές σε αυτή την επιτροπή έχω δει ότι, και έχω επιμείνει ότι η πληροφόρηση δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, πρέπει να απευθύνεται και προς τις επιχειρήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν γνωρίζουν ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτές οι επιχειρήσεις δηλαδή που επινοούν αυτές, αυτά τα προϊόντα ή τι υπηρεσιε πολλές φορές δεν έχουν κατά νου ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα και ανάγκες των καταναλωτών και μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ε, διαφορές, σε στη συνέχεια. Η επόμενη τροπολογία ε, για την παράγραφο 16 έχει κάποιες προτάσεις τροποποίησης για τον νέο αηφόρο τρόπο κατανάλωσης. Γιατί η κατανάλωση του αύριο στις χώρες μας, που ήδη είναι ιδιαίτερα καταναλωτικές, θα είναι διαφορετική ποιοτικά και ποσοτικά. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε ε, τις σπατάλες, να προωθήσουμε την ανακύκλωση Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τέλος. Όλα αυτά θα πρέπει να εντάσσονται και στο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 που είναι εξαιρετικά δύσκολο σημείο βεβαίως ε, ε, που φτύρει και τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων αλλά το σημείο 17 της έκθεσης ε, τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση κατάλληλη, αλλά και ε, επαρκώς φιλόδοξη θα τη χαρακτήριζα εγώ, γιατί είναι από τους ε, τομείς που λαμβάνεται μικρότερη χρηματοδότηση. Και να πω παρεμπιπτόντω ότι εκπλήσωμαι από πολλέ τροπολογίε συναδέλφων, ιδίω από το ΕΛ, και προτείνουν απλώ τη διαγραφή αυτή τη παραγράφου. Από πλευρά μου δεν θέλω να διαγραφεί. Θα ήταν ε, ένα κακό σημάδι, κακό μήνυμα στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου. Και ίσως να θεωρηθεί και ανεπαρκή σε στήριξη και προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ αγαπητέ φίλε. Ας πω λίγα λόγια ως σκιώδης εισηγητής για την πρόταση. Συνεργάστηκα με την κυρία Κανιέτη, Καρνιέτε μάλλον, γιατί έχουμε μερικά κοινά θέματα και ορισμένες τροπολογίε τροπολογίες που υπογράφουμε από κοινού. Και δώσαμε ιδιαίτερα βάρος σε μια απάντηση στην πρόταση της Κομισιόν, γιατί είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να στοχεύσει ιδιαίτερα στο να, δώσουμε, να βάλουμε προτεραιότητες και να προσφέρουμε και νέες ιδέες προτάσεις της Κομισιόν. Και είναι σημαντικό αυτό για τους καταναλωτές και για ορισμένες νέες τάσεις. χωρίς να προσθέσουμε νέα, νέους τομείς, εάν δεν είμαστε βέβαιοι ότι εντάσσονται πραγματικά στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγία. Το γεγονός ότι υπάρχουν τώρα τόσε πολλέ τροπολογίε, αυτό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουμε το ρόλο μας στα πλαίσια της προστασίας των καταναλωτών. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ω εξή μερικά σημαντικά πράγματα. Και τα σκέφτηκα εγώ και τα υποβάλλω στην προσοχή σας. πρέπει να επαγρυπνούμε περισσότερα για πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού για τους καταναλωτές, γιατί έχω κάπως την αίσθηση ότι δεν προσέχουμε αρκετά σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις έλλειψης ανταγωνισμού στους καταναλωτές. Ξέρω ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είχαν μάλιστα και μία μονάδα καταναλωτών, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή. Πάντως το θέτω αυτό το θέμα επίτηδες, διότι οι συνάδελφοί μας της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής ανησυχούν και δικαίως για θέματα γύρω από κανονισμούς ε, οικονομικών υπηρεσιών και την σταθεροποίηση του ευρώ. Και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν πολύ με την πολιτική ανταγωνισμού. Μίλησα με την Sharon Bowles και δεν διαφωνεί μαζί μου. Δεν είναι υψηλά στι προτεραιότητε του. Υπάρχουν και σημαντικέ υποθέσεις μια θεωρούμενη ω. θεωρούμενη, συγγνώμη, θεωρούμενης ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισμό συμπεριφοράς στον ψηφιακό κόσμο ιδίω. Όπου, για παράδειγμα, προτείνονται κάποιες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, αυτές να είναι πραγματικά ανεξάρτητες και να προσφέρουν πραγματικά μια υπηρεσία στους καταναλωτές, όχι να εξυπηρετούν αυτόν που την έχει φτιάξει. όποιο και να τι έρχεται στι ιστοσελίδε αυτές, να τι διαχειρίζεται κάποιο με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό, ώστε οι καταναλωτέ να μπορούν να βασιστούν σε αυτέ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα γίνει όλο και πιο δύσκολο και το οποίο διασυνδέεται επίση με την εργασία που γίνεται για προστασία δεδομένων και πώ χρησιμοποιούνται για, για, για το μάρκετινγκ τα δεδομένα των καταναλωτών. Έκανα και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με εκπρόσωπο των Βρετανών καταναλωτών και μου μιλούσε για τα συμφέροντα των καταναλωτών στον ψηφιακό χώρο και ότι έχουν εντοπίσει ορισμένες περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές ανάλογα με τις προφορίες του προφίλ τους λαμβάνουν διαφορετικές προσφορές από άλλους καταναλωτές ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους που προκύπτουν από την αναζήτηση που κάνουν στο διαδίκτυο. Είναι θέμα και η προστασία των καταναλωτών αυτό. Πρόκειται για νέε προκλήσεις τι οποίε τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και επειδή συνεχίζουμε τη δουλειά μας στην ψηφιακή ενιαία αγορά και τα όσα είπε ο κύριος Μπαρνιέ το πρωί, ότι θα θέλαμε να τα εντάξουμε σε μία πρωτοβουλία ενιαία για την ε, ενιαία αγορά, φέτος το φθινόπωρο, ίσως είναι σκόπιμο να παρακαλέσουμε τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και δικαιοσύνη. να μοιραστούν ορισμένε σκέψει μαζί μα που να μπορέσουμε να τι διοχετεύσουμε προ τα εκεί. Θέματα πολύ σημαντικά νομίζω για του καταναλωτέ στο μέλλον. Ο δεύτερο τομέα που συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και είναι μάλλον βασισμένο σε πληροφοριε information based. Νομίζω δηλαδή ότι δεν κάνουμε αρκετή χρήση των πληροφοριών και καλών πληροφοριών που συλλέγει η Γενική Διεύθυνση Σάρκο για τους καταναλωτές. Υπάρχει ένας πλούτος πληροφοριών, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι τη χρησιμοποιούμε σωστά. Θα κάνω μια πρόταση που ελπίζω να αποδειχθεί εφαρμόσιμη. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών προτείνει να κάνει κάποια εργασία για την οικοδόμηση κάποιων προτύπων για την ενιαία αγορά. Και θα γίνει και μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου δυστυχώς δεν μπορώ. Μάλιστα ήταν σήμερα η σε αυτή. Βεβαίως δεν μπορούσα να πάω γιατί είχαμε τις ψηφοφορίες το σημερινό πρωινό. Πάντως έγινε η συνάντηση αυτή για αυτό το λεγόμενο modeling work, δηλαδή η δημιουργία μοντέλων για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων των καταναλωτών. Πολλή δουλειά μπορεί να γίνει εκεί και νομίζω ότι θα βρει την θέση της η δουλειά αυτή μέσα στα πλαίσια αυτή της πρωτοβουλίας υπέρ των καταναλωτών. Να λοιπόν μερικέ σκέψεις που ήθελα να σας θέσω υπόψη και τελειώνοντα γιατί έχω και ορισμένε άλλε τροπολογίε άλλων συναδέλφων που έχω δει και που θεωρώ ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ορθή ροή πληροφοριών και ενημέρωση των καταναλωτών και ασφαλείας τους. Να, υπάρχει, να, να, δηλαδή να, ληφθούν οι αποφάσεις, το policy making να γίνεται βασισμένο σε επιστημονική θεμελίωση και εκεί εξυπηρετεί και η υποπτία των αγορών. Αυτά τα θέματα βέβαια είναι οριζόντια μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και είναι σημαντικό να καταστήσουμε σαφές γιατί το θεωρούμε αυτό σημαντικό. Ε, αυτά ήθελα να συνεισφέρω ως σκέψεις και επειδή η κυρία Ρίουλε δεν έχει έρθει ακόμη, νομίζω εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ε, ο κ. Κρότσμαν. Όχι, καλά λοιπόν. Μπορούμε ίσως να ζητήσουμε, αν συμφωνείτε εσείς κύριε Σιγητά, από την Κομισιόν. Κύριε Σπανού. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε και για τα πολύ καλά σας λόγια στην αρχή Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να είμαι σήμερα εδώ παρούσα. Σας γνωρίζω όλους πολύ καλά λόγω των προηγούμενων καθηκόντων μου και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Και ιδιαίτερα ξεκινώντα ε, με στα πλαίσια των καθηκόντων μου την ατζέντα των καταναλωτών, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε πολύ θετικά αυτό το έργο. Όλοι κινούμε προς τον ίδιο στόχο και εγώ προσβλέπω στις τελικές ε, να ολοκληρωθούν συζητήσεις και να έχουμε και τελική έκθεση. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης. Καταγράφουμε όλα τα σχόλια. Ένα σχόλιο για τους τροπολόγιους που έχουμε δει. Και ήδη σα έχουμε κάνει κάποιε πατρίδε και εμεί. Η κυρία Μανφρέντ είναι μαζί μου από την ΓΑΜΑ Δικαιοσύνη, όπω είπατε, Μάλκομ, γιατί είναι κοινή πρωτοβούλια. Και η Κομισιόν είναι ενιαία και η ατζέντα είναι ενιαία γιατί οι καταναλωτέ είναι παντού στην Ευρώπη, οπότε ανάλογα με την υπηρεσία που εστιάζει σε αυτούς κάθε φορά ο καταναλωτή, αλλάζει το πλαίσιο Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η προσφυγή. Η προσφυγή είναι στο μέσο στον οποίο συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Παραμένει στην ατζέντα, όχι μόνο και τώρα υπάρχει συμφωνία που υπήρξε πλέον το τελευταίο Δεκέμβρη ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τις εναλλακτικέ μεθόδους επίλυσης και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έτσι μπορούμε να διεκνούσουμε καλύτερα το αρχικό κείμενο για την προσφυγή σε ενδικά μέσα ώστε να είναι ξεκάθαρη η χρήση ε, των εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών όπως και τις, ε, των συλλογικών προσφύγων. Είναι και τα δύο μέσα, αλλά είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και χαίρομαι γιατί υπάρχει πλέον αυτή η συμφωνία πλέον για τα EDR-ODR. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ήδη υπάρχει δέσμευση μέσα στα πλαίσια του SMA2 και κάνουμε το follow-up της όλης διαδικασίας. Ήδη στο πρόγραμμα μας προβλέπεται ένα πακέτο να υιοθετηθεί για τη διαφάνεια πρόσφαση ε, και για την αλλαγή τραπεζικών λογαριασμών. Το δουλεύουμε αυτό το πακέτο, οπότε θα επανέλθουμε σύντομα. Και πάλι είναι σημαντικό η έκθεση να λάβει υπόψη και αυτό το στοιχείο και να μην παραγνωρίζει ότι ήδη έχουμε κάνει αξιολόγηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη και το μη ικανοποιητικο follow follow-up των αρχικών συστάσεών μας, οπότε ήδη α, είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία και συγκεκριμένη πρόταση με την ασφάλεια των προϊόντων. Και πάλι κινούνται τα πράγματα. Η ατζέντα των καταναλωτών είναι κάτι δυναμικό. Την προηγούμενη εβδομάδα υιοθετήσαμε ένα πακέτο για την εποπτεία τη αγορά και την ασφάλεια των προϊόντων. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να προκύψει ε, μέσω τροπολογιών για την προστασία της πηγής, προϊόντα δηλαδή από τέτοιες χώρες. Σίγουρα χρειάζεται συνεργασία με τρίτε χώρε. Δεν έχουμε την νομική βάση για να κάνουμε εμεί αυτέ τι επιθεωρήσει, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, το ότι οι επιθεωρήσει γίνονται από τι αρχέ των χρόνων αυτών. Τώρα για τι οργανώσει καταναλωτών. Πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να τι στηρίζουμε. Είναι η προσέγγιση μα αυτή. Του στηρίζουμε χρήματο, χρηματοδοτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με capacity building επίση. Δύσκολα βλέπουμε το θετικό ενό μητρώου για οργανώσει καταναλωτών θα πετύσει τεράστια δουλειά και δεν ξέρω τελικά αν θα μας δώσει τα επιδιωκόμενα. Σε ό,τι αφορά την ευαλωτότητα των καταναλωτών, στην ίδια κατεύθυνση με δική μας ε, πρόθεση, ιδιαίτερα ευάλωτος ορατής είναι μια, ένας γενικός όρος. Κινείται από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, οπότε ίσως είναι σκοπό να μην μιλάμε για ευάλωτους καταναλωτές, αλλά για ευάλωτες καταστάσεις ιδίω μέσα στα πλαίσια της κρίσης. Δουλεύουμε λοιπόν από αυτού, γίνονται μελέτες για αυτό το ζήτημα και εστιάζουμε σε αυτό το τομέα. Ποιότητα των προϊόντων με μάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός της νομοθεσίας μας είναι η ασφάλεια πάνω απ' όλα των τροφίμων και λοιπών προϊόντων. Όταν μιλάμε για ποιότητα, για τα τρόφιμα υπάρχει ειδική γεωργική νομοθεσία, αλλά για τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων και υλικών στις διάφορες αγορές. εκεί είναι θέμα α, συνηθιών, επιλογών του καταναλωτή. Και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη συζητήση για την ενέργεια που αναφέρεται και σε κάποιες τροπολογίες. Να σας πω ότι μετά την εντολή που λάβαμε από τον Φόρουμ, δημιουργήσαμε ε, μία ομάδα εργασίας ε, σχετικά με σκοπό την ε, ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενημέρωση του καταναλωτή σε θέματα ενέργειας και εκεί γίνεται λοιπόν δουλειά. Τώρα, για την ε, ανακοίνωση, για την επικοινωνία, συγγνώμη, για την επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία γίνεται μαζί με τα κρατημέλη. Ήδη κάνουμε μια εξάκτη αξιολόγηση για να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε κατάσταση ώστε από κοινού με τα κράτη-μέλη να βρούμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Σύγκριση τιμών. Χαίρομαι που το αναφέρατε και αυτό είναι πολύ σημαντικό Η σύνδεση κορυφή των ε, Ευρωπαίων Καταναλωτών λαμβάνει η χώρα την επόμενη εβδομάδα και εκεί προετοιμαζόμαστε να τοποθετηθούμε και αυτό το θέμα. Εκεί έχουμε τους ε, ενδιαφερομένους από πολλούς τομείς και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω με τα σχόλιά μου να βοηθούμε και εμείς. Και εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μανφρέντι θέλει το λόγο, παρακαλώ. Εν συντομία, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να επισημάνω πόσο και εμείς εσπαζόμαστε στις δικές σας θέσεις. Ότι δηλαδή θα πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία των ψηφιακών καινοτομιών και εξελίσσεων, την αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών βάσει τη Πραγματικά αυτή η οδηγία δημιουργεί ένα τεράστιο δυναμικό για να αντιμετωπίσουμε την κατάχρηση του ίντερνετ και της δυνατότητας να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Η Επιτροπή σας σύντομα θα λάβει μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας περί πρακτικών. Ελπίζουμε στα μέσα Μαρτίου, πριν και τη Σύνοδο Κορυφής για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή και όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που στηρίζουν την ουσία της ατζέντα αυτής. Ιδίως τι εννοώ. Σε μια εποχή περιορισμού των πόρων σε όλους τους τομείς, Μιλώ για περιορισμό οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Απεγνωσμένα λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις προτεραιότητες. Η ατζέντα αυτή τι κάνει λοιπόν. Επιλέγει πέντε οικονομικούς τομείς κλειδιά, όπου θεωρούμε ότι ελοχεύει κίνδυνο σημαντικός για τους καταναλωτές. Και βλέπουμε ότι σε μεγάλο βαθμό όλε τι τροπολογίε υποστηρίζουν την προσοχή μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ από τι Βρυξέλλε έχουμε περιορισμένε δυνατότητε. Πρέπει το Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει για να εστιάσουμε τι προσπάθειές μας. Τέλος, πολλά σημαντικά διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε από τέτοιες περιπτώσεις όπως η υπόθεση Μήλου που ίσως να την διαβάσα και σε εφημερίδες και αυτό που έγινε με την Επίτροπο Ρέντινγκ, η οποία και σε όλο του Υπουργό, λέγοντα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα κατάχρηση. Κατάχρηση που κάνουν οι έμποροι, που δεν λειτουργούν ξεκάθαρα διασνοριακά, αλλά ε, εντοπίζουν, στοχεύουν πολλούς καταναλωτές σε πολλές εσωτερικές εθνικές αγορές. Παίρνουμε σε νέες εποχές. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρία που μας δίνει η πολιτική ανταγωνισμού και να ορίσουμε κάποια κοινωτικά κατόφλια για υποθέσεις όπου απαιτείται μια πιο ισχυρή αντίδραση και πιο ισχυρή εφαρμογή στο Μόνο με τη στήριξη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Um, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε και για τις ε, φρέσκες ιδέες που μας δώσατε γύρω από το ίδιο θέμα. Ελπίζουμε πραγματικά σε αυτή η έκθεση να βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η οδηγία για τις αθέμενε πρακτικές ήταν πολύ σημαντική στην και ήταν κάτι που ε, μας μα απασχόλησε και μας παραπολιτώσε το λόγο στον εισηγητή να συνοψίσει αν θέλει την συζήτηση. Μας επιβεβαιώσατε το χρονοδιάγραμμα ούτως ή άλλως. παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και για τη δουλειά που έκαναν και τις προσπάθειες που έχουν κάνει για να έχουμε ένα καλύτερο τελικό κείμενο. Ευχαριστούμε και την ε, Επιτροπή για την αρχική προσπάθεια που κινητοποίησε την όλη διαδικασία, όπως και τις προτάσεις που ακούστηκαν και σήμερα στη συζήτηση. Ακολουθώντας βεβαίως ε, την ίδια γραμμή με όπως προηγούμενες συνεδριάσεις. Η έκθεση αυτή για την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική, γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλεγόμαστε, είμαστε επιλογή των ε, πολιτών και ε, από αυτούς εξαρτώμεθα και εν προκειμένου μιλάμε για τους πολίτες καταναλωτές, για τη δημιουργία του δουλειού του καταναλωτή. Και για μας ο πολίτης καταναλωτής είναι το επίκεντρο της πρωτοβουλίας. Είναι αρχή και το τέλος ε, αυτής της εργασίας. Στην πρώτη της έκθεση που μας έστειλε η Κομισιόν, έπρεπε να κάνει μια θετική διακρίση ανάμεσα ε, στην εγκάρσια προσέγγιση αυτής ε, της ε, πρότασης, κάτι που για μας είναι η βάση των εργασιών μας. Οι προτάσεις που έκανε αδελφή με στροπολογιών, ήδη περιλαμβάνονται, θα έλεγα, οι πλέον σημαντικές και τις ασπάζουμε και τις ημερίζουμε. Αναφέρουμε στροπολογίες εκείνες που μιλούν για περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της ικανότητας του καταναλωτή να ασκήσει τα καθήκοντά του σε μία όχι παρατηφιλική αγορά. Με αναγκαιότητα να έχουμε πιο καλούς μηχανισμούς και εργαλεία, ώστε οι πληροφορίες να ρέουν με τον καλύτερο τρόπο. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που ήδη έχουμε, αλλά βάζοντα και καινούριου μηχανισμού στο τραπέζι, γιατί υπάρχουν και νέε προκλήσει που αντιμετωπίζει ο καταναλωτή. Ό,τι κινείται γύρω από το εμπόριο, ό,τι κινείται γύρω από τι νέε τεχνολογίε, γύρω από την ανατεχνολογία, του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, όλε αυτέ τι πτυχέ τη τεχνολογική εξέλιξη, είναι στοιχεία που θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον καταναλωτή και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή την ατζέντα. Επιμένω λοιπόν στην ε, επικείμενη συνεδρία με τους Κιώδης να κάνουμε μία καλή δουλειά για να φτάσουμε σε μία συμφωνία για τα πλέον σημαντικά συστήματα. έχω και έναν κατάλογο σημαντικών τροπολογιών που θα προτείνω, θα τις λάβετε και γραπτός. Και ευελπιστώ ότι πραγματικά είμαστε στις κατάλληλες τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να προτείνουμε ουσιαστικές ε, συμβαστικές τροπολογίες στην Κομισιόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα το ανέφερα πριν. Θέλετε να το επαναλάβω. Όχι, έτσι. Μπορείτε να επενθυμίσετε αν θέλετε εσείς μόνο τις ημερομηνίες. Anyway έτσι κι αλλιώς θα δημοσιευθούν στον ιστοτόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρθές, που ηγηθήκατε αυτού του εγχειρήματο και προς όλους τους χειώδες. Σίγουρα η έκθεση θα είναι πολύ καλή. Ευχαριστούμε πολύ και την Επιτροπή για τις ε, παρεμβάσεις της. Μπορούμε να περάσουμε... Α, συγγνώμη, κυρία Καρνετή. Ευχαριστώ. Δράτω με τις για να απαντήσω στον κύριο Ροσφόρ, γιατί το ΕΛΚ πρότεινε τη διαγραφή στην αναφορά στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διαγράψαμε την παράγραφο 17, μιλάμε για την τροπολογία 208, γιατί έχουμε συμπεριλάβει ακριβώς αυτή την έννοια στην παράγραφο 5, τροπολογία 124. Βεβαίως, και το ΕΛΚ είναι απολύτως πεπισμένο ότι υπάρχει ανάγκη για έναν ε, επαρκή προπολογισμό για όλες αυτές τις ενέργειες. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι ικανοποιήσατε και την περιέργεια του κύριου Ροσφόρ. Εντάξει, περάσουμε στο επόμενο σημείο. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για μια σημαντική γνωμοδότηση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. θεωρούμε την εσωτερική αγορά ω ε, βασική προτεραιότητα τη Επιτροπής μα. Δεν είναι καθήλυνα αρμόδια δική μας ε, η Επιτροπή μα. Παρ' όλα αυτά, μαζί με την Επιτροπή Βιομηχανία, έχουμε καταλήξει μια συμφωνία για συγκεκριμένα σημαντικά στοιχεία. Η κυρία Κάλλα, λοιπόν, έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για αυτό το πακέτο και ξέρω ότι Ήδη και κάποιες συναντήσεις ε, με τον κλάδο. Κυρία Γκάλα, θα σας δώσω το λόγο γιατί είναι η πρώτη ευκαιρία που έχετε για να μας παρουσιάσετε αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν είχατε προετοιμάσει κάτι για την αξιολόγηση αντικτύπου που έχετε ζητήσει από την Επιτροπή. Είναι εδώ όμως η Επιτροπή, όπως και να έχει. Αντρέα Σαββίδιος, είστε εδώ. Ωραία. Είναι επικεφαλής ε, της ε, Task Force στην Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκάλο πρώτα απ' όλα. Και μετά από ό,τι κατάλαβα η Επιτροπή θα μας ε, παρουσιάσει την πρόταση. Παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο, αλλά και ιδιαίτερα τεχνικό. Έχω λοιπόν κάποια ερωτήματα να απευθύνω προς ε, την Επιτροπή. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνετε το λόγο πρώτη. Αυτή η πρόταση κανονισμού συμπεριλαμβάνει νέα, σημαντικά νέα στοιχεία καινοτομία, γιατί σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή οδηγία του 1999, αυτή η πρόταση πέραν της ηλεκτρονικής υπογραφής εισαγάγει νέες ε, υπηρεσίες εμπιστοσύνης όπως ε, η σφραγίδα ε, και αναφέρεται και στην, στο παραδεκτό κάποιων ηλεκτρονικών εγγράφων και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης τέτοιων εγγράφων. Θεωρώ ότι είναι σημαντική και η επιλογή του κανονισμού. Στηρίζω την επιλογή αυτή της Επιτροπής γιατί πράγματι η οδηγία του 1999 δεν είχε τις ε, αναμενόμενες ε, επιπτώσεις ό,τι φορά την εναρμόνιση. Η εφαρμογή ε, ποικίλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος εξαιτίας διαφορετικών ερμηνεών από τα κράτη-μέλη. Φάνηκε ότι υπήρχαν προβλήματα διαλειτουργικότητας και βεβαίως κάτι που ξέρουμε και μας λυπεί παρατηρείται και ο κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς. Πέραν αυτού, τα πρότυπα της οδηγίας του 1999 ε, θεωρούνται πλέον παροχημένα σε σχέση με τις ε, προσδοκίες της αγοράς. Στο όχι αυτής της ε, πρότασης κανονισμού είναι σαφής και δεν απέχουμε εδώ και από το ζήτημα που μας απασχόλησε προηγουμένως, δηλαδή η δημιουργία όρων και προποθέσεων εμπιστοσύνης ε, για τους καταναλωτές και βεβαίως ένα τέτοιο ψηφιακό περιβάλλον είναι κάτι σημαντικό και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή την ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτή η όρη εμπιστοσύνη ε, σίγουρα εξαρτώνται και από την τήρηση ε, και το σεβασμό μάλλον των προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο θέμα είναι και αυτό ένα ζήτημα που γνωρίζω καλά. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί λοιπόν. Ιδίω εφόσον αυτό ο κανονισμός θα πρέπει να συνάδει και με τα όσα κάνουμε εμείς τουλάχιστον στη Γιούρη σε ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον ιδιωτικό βίο. Privacy by design. Σημαντικό σημείο για μας αυτό. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της, ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς, εμείς καλούμε και πάλι προς την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά δυστυχώς δεν τον έχουμε επιτύχει ακόμα. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία για τα οποία μου ετέθησαν κάποια ερωτήματα, ή μάλλον εγώ θέτω κάποια ερωτήματα και θα ήθελα τις εξηγήσεις ε, της ε, Επιτροπής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την αρχή της, ανα... της και της ε, παραδοχή ε, παραδοχής ε, που έχει εισαγάγει η Επιτροπή, είναι μια καλή επιλογή, εφόσον επιτρέπει σε κάθε κράτο μέλος που έχει ήδη επενδύσει και αναπτύξει τέτοια μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, να τα διατηρήσουν τα συστήματά τους. Ωστόσο, η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών είναι σημείο κλειδί για την ανάπτυξη του ψηφιακού περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο αυτό το σύστημα κοινοποίηση που προτείνεται θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκές ε, σε σχέση με τα πρότυπα ασφαλείας που προτείνονται. Έτσι, το ερώτημα που θέτω εγώ είναι πρέπει να εισαγάγουμε προδιαγραφές και ελάχιστα κοινά πρότυπα όπως αυτά που έχει ε, προτείνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτύπων ε, Ταυτοποίησης. Υπάρχουν ήδη κάποια τέτοια πρότυπα που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς, δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί, αλλά μας επιτρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο σημείο αναφοράς. Δεύτερο σημείο που με απασχολεί αφορά την ε, ταυτοποίηση για τις νέες υπηρεσίες εμπιστοσύνης ε, που έχουν εισαχθεί ε, σε ό,τι φορά τη σφραγίδα και τα ηλεκτρονικά Εδώ μιλάμε για την αμοιβή αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών και τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της νομικής ασφάλειας. Μια πολιτική ε, πιστοποίησης λοιπόν που επιφέρει ενιαία νομική ερμηνεία. Για μένα είναι ένα, πολύ ουσιαστικό σημείο αυτή τη πρόταση ό,τι φορά την, ε, και την χρήση τέτοιων υπηρεσιών εμπιστοσύνη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και βεβαίω υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ε, κανονιστικού πλαισίου για τις ε, δημόσιες προμήθειες, ε, για την ανάπτυξη του e-procurement, το είχαμε θίξει αυτό το θέμα και εδώ πλέον πρέπει να περάσουμε στις πράξεις και να μην μένουμε μόνο στα λόγια. Τρίτο σημείο προβληματισμού αφορά τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, δηλαδή άρθρο 17 παράγραφος 1. Και εδώ το ζήτημα είναι η έλλειψη υποχρέωσης ε, απόκτησης πρώτερης άδειας πριν δηλαδή την παροχή των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, εάν ε, η έκθεση ελέγχου που δίνεται σε αυτό το όργανο ελέγχου αποδεικνύεται ότι δεν έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, τι συμβαίνει. Εδώ θα ήθελα η Επιτροπή να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Άλλο στοιχείο, Πενθυμίζω ότι στο ψήφισμα της 16ης Ιουνίου 2010 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει μια πύλη ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ στο σημείο 26 η Επιτροπή έχει θεσπίσει αυτές τις υπηρεσίες έγκρισης, αλλά δεν λέει ποιος ακριβώς θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Υπηρεσίες έγκρισης απαλήθευσης Και εδώ θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Τέλος, ακόμα και αν κατανοώ ότι δεν μπορούμε τουλάχιστον σε αυτή την Επιτροπή να συζητούμε επάπειρον τις τεχνικές προδιαγραφές. Η τεχνολογική ουδετερότητα επιβάλλεται σε αυτή την πρόταση, όμως θεωρώ ότι η συστηματική προσφυγή στις ε, κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις είναι υπερβολικά τακτική και συστηματική. Θα πρέπει να διορθωθεί αυτό μέσω προτάσεων της ε, Επιτροπής. Οφείλει να υποβάλλει τις προτάσεις της Επιτροπής, λοιπόν. Κλείνω αυτή την αρχική παρουσίαση. παραπέμποντας και ε, στην ε, σύγκρουση συμφερόντων που έχουμε και αρμοδιοτήτων που έχουμε εδώ πέρα στο, σε αυτό το φάκελο. Αυτή η πρόταση αρχικά ανατέθηκε στην Ήτρε. Ο πρόεδρος μας ε, πολύ καλά έκανε και διαμαρτυρήθηκε γιατί θεωρώ ότι η ψηφιακή εστερική αγορά είναι δική μας αρμοδιότητα Πολλά υπόθηκαν στη συνδιάσκεψη των ε, Προέδρων και φτάσαμε μέχρι και το άρθρο 51 μεταξύ της Ήτρε και της Γιούρη. Έχουμε ένα άρθρο 50 με την ε, Επιτροπή Ήτρε και μετά από αυτές τις ε, μακραίες και δύσκολες διαπραγματεύσεις θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι να στηρίξουμε αυτή την πρόταση και ελπίζω και οι σκιώδεις εισηγητές να συμφωνήσουν μαζί μου. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο Χάρμπουρ που πολύ επιτυχημένα περασπίστηκε τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Και πάλι περιμένω τις εξηγήσεις της Επιτροπής γιατί πράγματι είναι ιδιαίτερα τεχνικό αυτό το θέμα Χαίρομαι τουλάχιστον που βρίσκονται όσοι συνάδελφοι κατάφεραν να βρεθούν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ που περιγράψατε τα πιο κρίσιμα σημεία. Έχετε βέβαια και την εμπειρία στα θέματα αυτά και ευτυχώς που υγείστε εσείς της προσπαθίας. Δύο σκιώδεις, Πρέντεργκαστ και εγώ προσωπικά. Α, Κρότσπαν επίσης. Α, ναι, ναι, ναι, αντικαθοστάτε τον κύριο Μπουσόη. Έχουμε λοιπόν και έναν αναπληρωτή σκιώδη συγητή. Θα παρακαλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να προβεί στην ε, τοποθέτηση από πλευρά της Κομισιόν. Να ακούσουμε λοιπόν εσάς αγαπητέ κύριε στο πλαίσιο των παρατηρήσεων της κυρίας Γκάλο και μετά ας αρχίσει με τις ερωτήσεις η κυρία Πρέντεργκαστ που θα την ακολουθήσει ο κύριος Κρότσμαν και μετά εγώ και εν τέλει θα μας εξηγήσει το χρονοδιάγραμμα η κυρία Γκάλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Συγήτρια και καλησπέρα σε όλες και όλους. Μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να παρουσιάσω την πρόταση. Θα προσπαθήσω μέσω της παρουσιάσεως αυτής να σας προσφέρω ορισμένε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσε η εισηγήτρια. Και στο τέλος της παρουσιάσεως ίσως μπορώ με τις ερωτήσεις και απαντήσεις να μπορέσω να ολοκληρώσω. Γιατί λοιπόν κανονισμός. Η εισηγήτρια εξήγησε δύο θέματα, τον κατακαιρματισμό πρώτον που προέκυψε από την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή και δεύτερο σημαντικό, με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε σχέση με την ίδια την πρόταση τις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν σε ορισμένες χώρες μέλη για να γίνει η ηλεκτρονική υπογραφή, το πλαίσιο δηλαδή αυτό και οι τεχνικές δυνατότητες να μπορέσουν να λειτουργήσουν στο εθνικό επίπεδο. Η Οδηγία 99 δεν φτιάχτηκε για να προσφέρει τα ειδικά εργαλεία για την ανάπτυξη, την εθνική ανάπτυξη, αλλά να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας αγοράς και η ηλεκτρονική υπογραφή να αποτελέσει ένα βήμα δημιουργίας εμπιστοσύνης, να αυξηθεί το επίπεδο αξιοπιστίας. Αυτό δυστυχώς δεν συνέβη και πιστεύουμε ότι αφενός η επιλογή του εργαλείου, δηλαδή κανονισμός, είναι πράγματι ο σωστός τρόπος για να μπορέσουμε να υπερβούμε τους κατακαιρματισμούς που μας έπληξαν σε σχέση με την ηλεκτρονική υπογραφή. Δεύτερη πτυχή. Η οδηγία εγκρίθηκε το 1999. Πέρασε πολύ καιρό από τότε και δεν μιλούμε πλέον για υπογραφή, μιλούμε για trust services, υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ένα σημαντικό θέμα στο ψηφιακό πλαίσιο είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα επιτρέψει ταυτοποίηση. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι μόλις θίξουμε το θέμα της ταυτοποίησης μπαίνουμε σε πολύ ευαίσθητο έδαφος. Το να δώσει κανείς ε, την ταυτοποίηση είναι αρμοδιότητα χωρών μελών. Με τον κανονισμό δεν επιβάλλουμε ένα αρμονισμένο πλαίσιο είτε για ταυτοποίηση είτε για ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ανοίγουμε δρόμους, προσφέρουμε δυνατότητες γιατί πάνω από 16 χώρες μέλη ήδη εξελίσσουν κάποιου είδους ηλεκτρονικά μέσα ταυτοποιήσεως για τους πολίτες τους ώστε να μπορούν αυτοί να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες επιγραμμικά και εμείς θέλουμε τώρα από αυτό να μπορεί να επεκταθεί και εκτός ε, πλαισίου αρμοδιότητας. Εκτός δικαιοδοσίας μάλλον να το πω πιο σωστά. Επομένως η αμοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών εμπιστοσύνης και μέσων ηλεκτρονικής ε, ταυτότητας για να επιτραπεί η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη βάση του άρθρου 114 και να ενταχθεί στο πακέτο του νομικού πλαισίου που πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί για να ενισχυθεί η ψηφιακή εμπιστοσύνη και να βασίζονται οι πολίτες σε τέτοιες υπηρεσίες, σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Όπως λέχθηκε από την εισηγήτρια, έχουμε κάνει ένα βήμα ή ορισμένα βήματα μπροστά μετά από την οδηγία της ηλεκτρονικής υπογραφής. Προσπαθήσαμε να εναγκαλιστούμε και τα όσα προέκυψαν ως ανάγκες ή τα νομικά πλαίσια των χωρών μελών όπου ήταν γνωστό δηλαδή ότι η ίδια ηλεκτρονική υπογραφή ως τέτοια είναι σημαντική, αλλά αν θέλετε να την εφαρμόσετε πλησιάζει πολύ περισσότερο σε αυτά που χρειάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορέσουν πραγματικά να επωφεληθούν από τη διαδικασία αφιλοποίησης. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερα πράγματα και Βάλαμε και το time stamping, η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν τα όσα ήδη γίνονται στις χώρες μέλη να αναγνωριστούν νομικά και πέραν της μεθορίου. Και το ηλεκτρονικό έγγραφο που είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει θα καταστεί δυνατή η αφιλοποίηση, αποϊλοποίηση αν θέλετε. Θα είναι βέβαια δύσκολο να γίνουν αυτά τα πράγματα αν δεν υπάρχει κάποια ασφάλεια δικαίου και κυρίως μεταξύ επιχειρήσεων, business to business, αλλά και επιχειρήσεις με, και κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις και πολίτες. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι ο συνομιλητής μας, ποια είναι η ε, άλλη πλευρά, αν, αν πρόκειται δηλαδή για μια ιστοσελίδα και πώς συνδέεται με μια αληθινή οντότητα, με ένα πρόσωπο. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη διευκόλυνση, μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερες διαδικασίες που θα επιτρέψουν μακρόθεν ε, καταχώρηση για παράδειγμα χωρίς να χρειαστεί να πάει κανείς επί τόπου και χωρίς άλλα μέτρα ταυτοποίησης ή που μπορεί να είναι ήδη στα χέρια κάποιου πολίτου ή χρήστου και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον από τη τεχνολογική πτυχή και σε άλλες χώρες μέλη. Αλλά μπορεί να υπάρχουν αυτά τεχνολογικά μένα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η νομική αναγνώριση. Και εκεί πρέπει να καλυφθεί το κενό αυτό. Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις. Εάν έχετε μια επιχείρηση σε μια χώρα και θέλετε να μπορείτε να έρθετε σε επαφή και να συναλλαγείτε όχι μόνο με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και με όλο τον κόσμο. Αυτά είναι το πρώτο βήμα. Αν θέλετε να φτιάξετε λοιπόν ένα αξιόπιστο περιβάλλον το οποίο να διέπεται από ασφάλεια δικαίου, από accountability, από ασφάλεια και να διευκολυνθείτε, αυτά θα πρέπει να γίνουν βέβαια το στάνταρτ και στο διεθνές επίπεδο. Και αυτό ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, που αυτό για μας είναι μεγάλος στόχος της απελευθέρωσης, γιατί αυτές είναι ο η κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη. Στις επόμενες δύο διαφάνειες δεν θα επεκταθώ πολύ, ήθελα μόνο να διευκρινίσω γιατί πιστεύουμε θα καρποφορήσουν όλα αυτά τα μέσα υπέρ κάποιου ο οποίος θέλει να υποφεληθεί από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Βεβαίως ο φορολογούμενος Μπορεί να μην είναι και η καλύτερη δραστηριότητα του κόσμου, αλλά παρόλα αυτά και για αυτού, που είναι ίσω μια οδυνηρή διαδικασία πρέπει ωστόσο να γίνει ευκολότερη και ε, ελέγξιμη και αξιόπιστη. Γι' αυτό βλέπετε στα βήματα της ε, πρώτης διαφάνειας βλέπετε ποιο, ποια είναι η ψηφιακή πύλη, ποια είναι η διοικητική διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί και όταν γίνουν αυτά ίσως χρειάζεται να ταυτοποιηθείτε. Και γιατί κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται η ίδια διαδικασία. Σήμερα είναι για τα φορολογικά, αύριο θα είναι ίσως για να καταχωριστείτε σε κάποια άλλη υπηρεσία. Γιατί να έχετε διαφορετικά token, διαφορετικά σύμβολα, ας πούμε έτσι. Και όταν θα είμαι έτοιμος πλέον να υποβάλω τα έγγραφά μου, πρέπει να μπορώ να είμαι βέβαιος ότι αυτά που διαβιβάζω είναι πραγματικά αυτά τα σωστά που πρέπει να διαβάσω. Η υπογραφή βέβαια δεν σημαίνει απλά συγκατάθεση εκ μέρου μου, αλλά και ένα είδος φραγίδας που σημαίνει ότι αυτά που θα λάβει η άλλη πλευρά δεν θα μπορέσουν πλέον να ε, τροποποιηθούν, να παραχαραχθούν ή να αρνηθούν ότι τα έλαβαν. Βέβαια, εφόσον έχω κάνει εγώ την ε, το δικό μου καθήκον, πρέπει να λάβω κάποια απάντηση και από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό έχουμε εδώ το time stamping, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Μίλησε για το e-procurement η συγγετρία. Πρέπει λοιπόν μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται να μπορεί να υποβάλει την προσφορά της ε, στο κατάλληλο, χρονικό, ε, στο κατάλληλο χρόνο και επομένως να λάβει τη σχετική βεβαίωση. Και όταν θα τα έχετε κάνει όλα αυτά, βέβαια, να μπορείτε να τα διατηρήσετε όλα αυτά τα έγγραφα, ώστε να μπορείτε και αργότερα να αποδείξετε ποιες υπήρξαν οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας ή και αν κάτι συμβεί στο μέλλον να μπορείτε να αποδείξετε ότι τα όσα έχετε διατηρήσει ήταν ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι όπως έγινε δηλαδή στην ε, συναλλαγή. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για όλους τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις κυβερνήσεις και νομίζουμε ότι αυτά θα διευκολύνουν τη ζωή όλων, ιδίως των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά θα προσφέρουν και μια καλύτερη δυνατότητα οργάνωσης των διοικητικών διαδικασιών και επομένως να απλοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ε, δημόσια διοίκηση ή τέλος πάντων στο γραφειοκρατικό πλαίσιο. Το άρθρο τώρα, τα άρθρα τώρα που προσφέρουν αποκλειστική αρμοδιότητα στην Επιτροπή. Εμείς πιστεύουμε ότι η δέσμη αυτή πρέπει να εξεταστεί στο σύνολό της και χαιρόμαστε που ακούσαμε από την εισηγήτρια αναφορά και σε άλλα μέρη που ενδεχομένως δεν είναι εμπίπτωση στην αποκλειστική αρμόδιότητα της ΣΥΜΚΟ, αλλά χρειάζεται να εξασφαλιστεί η νομική ασφάλεια. Όπως είπα, ε, αξιόπιστα συστήματα, πιστοποίηση των προϊόντων και βέβαια την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εν προκειμένου θεωρούμε ότι ο κανονισμός βάζει κάποιες, βάσιμες, κάποιες ε, βασικές συγγνώμη, ε, απαιτήσεις με τον τρόπο βέβαια που θα υλοποιηθούν και τεχνολογικά οι απαιτήσει αυτές και οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε προδιαγραφές, στις εφαρμοστικές πράξεις δηλαδή, και που έχουν ως στόχο να υπάρξουν διαθέσιμες οι προδιαγραφές για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού. Επειδή βέβαια μιλούμε για υπηρεσίες που ακόμα δεν έχουν βρει ευρία διάδοση σε όλες τις χώρες μέλη, ίσως να μην υπάρχουν ακόμα έτοιμες οι σχετικές προδιαγραφές. Και γι' αυτό ή τα πρότυπα. Και γι' αυτό όταν θα υπάρξουν τα πρότυπα θέλουμε να υπάρχει ένας εύκαμπτος μηχανισμός, όπως άλλωστε έχουμε περιλάβει και σε άλλα νομοθετικά κείμενα, όπως στην οδηγία ηλεκτρονικής υπογραφής, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αναβαθμίζονται τουλάχιστον τα πρότυπα εκείνα τα οποία θα προσφέρουν τη δυνατότητα νομικής συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονισμού. Βασικός πυλώνας αλλά και βασική περιπλοκή στα πακέτα η αμοιβαία αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Αυτό όχι μόνο είναι απόλυτα σημαντικό για την πιστοποίηση των χρηστών, αλλά και των νομικών προσώπων, αλλά έχει σχέση και με το πώς προσφέρονται τα μέσα αυτά στο εθνικό επίπεδο. Δεν έχουμε αρμοδιότητες για να επιβάλλουμε νομικά πρότυπα ή πρότυπα ασφάλειας για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελίξουν οι χώρες μέλη τα προγράμματά τους ηλεκτρονικής ταυτότητας ή αναγνώρισης. Από την άλλη μεριά έχουμε διάταξη που με κάποιο τρόπο υποστηρίζει την, την νομική αναγνώριση τέτοιων μέσων και ο μηχανισμός συνεργασίας που θα επιτρέψει στις χώρες μέλη ε, να καθίσουν και να ορίσουν από κοινού όπως έγινε και σε τεχνολογικά έργα όπως η ΣΤΟΑ, να έχουν τη δυνατότητα να θεμελιώσουν τη τεχνολογική διαλειτουργικότητα και το σύστημα που θα προκύψει από την εφαρμογή του κανονισμού. Τώρα, για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ήθελα μόνο να σας δώσω έτσι μια στιγμή φωτογραφία των βασικότερων έχοντα ξεκινήσει από την ηλεκτρονική υπογραφή προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τις διατυπώσεις αλλά και να τις κάνουμε ακριβέστερες. Ποιο είναι το ελάχιστο δηλαδή σύνολο απαιτήσεων για την νομική αναγνώριση πέραν της μεθορίου γιατί δεν θέλουμε να ενισχύσουμε τον ισιωτικό χαρακτήρα ας πούμε, των εισαγωγικών που έχουμε ήδη αλλά αυτό που θέλουμε είναι, αυτό που υπάρχει δηλαδή στο εθνικό επίπεδο, να μην χρειάζεται να αλλάξει, εκτός πια και αν δεν είναι συμβατό με το περιεχόμενο του κανονισμού. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ορισμένες φορές ακούμε ότι ναι θα υπάρξει ένα νομικό κενό μετά από την υιοθέτηση του κανονισμού. Διόλου δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η διατύπωση του κανονισμού θα υπερισχύει απέναντι στις εθνικές νομοθεσίες που ίσως προβλέπουν διαφορετικά πράγματα, ιδίως για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και που αυτό θα οφείλεται στον κατακαιρματισμό που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία 14 χρόνια. Το άρθρο 10 τώρα, βεβαίως για μας η ανώτατη επιταγή είναι η, ηλεκτρονική ενιαία αγορά, αλλά θέλουμε να διευκολυνθεί και η παροχή υπηρεσιών. Και το περιβάλλον που λειτουργούμε είναι παγκόσμιο. Και όταν μιλούμε για πιστοποιημένους ε, παρόχους υπηρεσιών, έχουμε ένα είδος αναγνώρισης το οποίο θα επιτρέψει όχι μόνο στην Ευρώπη να αναγνωρίζεται το τι συμβαίνει εκτός Ευρώπης, αλλά και πιο σημαντικό, και εδώ μπαίνει το στοιχείο της αμοιβότητας, να έχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να αναγνωριστούν αυτά δηλαδή, στη βάση της αμοιβότητας και από τους απ' έξω. Για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, εδώ απλουστεύσαμε τις διαδικασίες, ή τις διατάξεις μάλλον, για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ώστε αυτές να αφορούν μόνο φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά πρόσωπα, γιατί για τα νομικά πρόσωπα έχουμε τις ηλεκτρονικές σφραγίδες που είναι καταλληλότερες, γιατί το νομικό πρόσωπο υπογράφει είτε μέσω ενός φυσικού προσώπου, είτε εφόσον δρά ως νομικό πρόσωπο, το μόνο που κάνει είναι να βεβαιώνει την προέλευση ή την αυθεντικότητα του σχετικού εγγράφου. Για τα νομικά αποτελέσματα των ηλεκτρονικών σφραγίδων. Εξήγησα για ποιο λόγο δρά και πώς δρά το νομικό πρόσωπο και για ποιο λόγο επιλέγεται εκεί η ηλεκτρονική σφραγίδα για να διασφαλίζεται, όπως είπα, η προέλευση και η αυθεντικότητα. Τίποτα δεν θα γίνει όμως εάν δεν καθορίζεται ο χρόνος. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό στο ψηφιακό πλαίσιο χρειάζονται κανόνες, καθιερωμένοι κανόνες και ιδίως σε ό,τι αφορά τη νομική αξία της χρονοσφραγίδα. για το εάν το έγγραφο ή η αίτηση ή οτιδήποτε άλλο έχει όντως υποβληθεί εγκαίρως και αν εκπληρούνται η υποχρέωση που προκύπτει από ε, το κείμενο του νόμου. Το ηλεκτρονικό έγγραφο είναι πολύ σημαντικό σε πολύ σημαντική συνιστόσα, όπως και η ηλεκτρονική παροχή. Η ηλεκτρονική αποστολή και παραλαβή του κειμένου. Να βεβαιωθεί δηλαδή ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο θα έχει την ίδια νομική βάση, την ίδια νομική αξία μάλλον όπως το έγγραφο πάνω σε χαρτί δηλαδή. Διότι θα υπάρξει νομικό κενό καθώς περνούμε από μια δικαιοδοσία σε άλλη. Βάζοντας όμως ένα πλαίσιο κανόνων θα ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και τις δημόσιες διοικήσεις να βασίζονται σε αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν σημαντικές διευκολύνσεις και που όπως είπα πρέπει να είναι αξιόπιστες. Νομίζω ότι μάλλον κάλυψα τις ερωτήσεις της ε, εισηγητρίας εκτός από την τεχνολογική ουδετερότητα που για μας είναι ο πυρήνας και γι' αυτό έχουμε και τις εφαρμοστικές πράξεις για να μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη ποια είναι τα πρότυπα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της οδηγίας ηλεκτρονικής υπογραφής ο μοναδικός έλεγχος στις ηλεκτρονικές υπογραφής οδήγησε σε ορισμένες χώρες στην δημιουργία ενός είδους μόνο μιας λύσης βασισμένη στο λεγόμενο hardware, δηλαδή μια εφιούς κάρτας ας πούμε, από την άλλη μεριά είχε υποχρέωση ο πάροχος να υπογράφει τις ε, ε, παροχές υπηρεσιών και οι δύο μπορεί να είναι αξιόπιστε, ε, οι δύο αυτέ οι δυνατότητε μπορεί να είναι αξιόπιστε, εάν, εάν βασίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα. Αλλά έχουμε τώρα και τι καινούργιε εξελίξει, cloud signing και ούτω καθεξή, που πρέπει και αυτέ να καλυφθούν ή να υποστηριχθούν από την νομοθεσία. Τέλο, για το πιστοποιητικό ασφάλεια, το οποίο επίση εφήγει δεν υπάρχει επίσημη νομική αμοιβαία αναγνώριση, συμφωνία τέτοια δηλαδή, μεταξύ χωρών μελών για την αμοιβαία αναγνώριση της πιστοποίησης ασφάλειας. Υπάρχουν μόνο συμφωνίες μεταξύ αρμοδίων αρχών. Επτά χωρών μόνο. Εν προκειμένου συζήτηση είναι σημαντική γιατί πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η πιστοποίηση ασφαλείας ένα πραγματικό στοιχείο του ενεργητικού για την βελτίωση της αξιοπιστίας των διαφόρων μηχανισμών. Ταυτόχρονα, ας μην δυσμονούμε ότι δεν διαθέτουν όλες οι χώρες μέλη τα απαραίτητα για να μπορούν να παράγουν ή να λαμβάνουν τέτοια πιστοποιητικά. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε με τις χώρες μέλη. Uh, Ευχαριστούμε για την τόσο εξαντλητική και πλήρη αυτή παρουσίαση. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση. Πρέπει να τη δούμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή. Πολύ ορθά είπατε ότι είναι πόσο σημαντική πρόταση για να μπορέσει να σταθεί με επιτυχία η όλη προσπάθεια για την ηλεκτρονική αγορά. Και είναι πολύ σημαντικό για μας καθώς σε εμπορικές συναλλαγές όπως ηλεκτρονικές προμήθειες. Υπάρχει οδηγία για τις μας προμήθειες που λειτουργεί τη στιγμή και υπάρχουν σε κάθαρα στοιχεία. Και εδώ έχουμε μια πρόταση που έρθει να συμπληρώσει κάποια κένα. Πρέπει λοιπόν να υιοθετηθεί και εγκαίρος. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά θα μπορεί να ξεκονομηθεί πολύς χρόνος από την επικύρωση εγγράφων. Και θα λέγατε γενικότερα Άλλες παρόμοιες προτάσεις όπως επί επαγγελματικές κάρτες, ηλεκτρονικές κάρτες συνδέονται άρρηκτα και με αυτή την ιδέα. Είμαστε... Ε, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να προχωρήσει αυτή η πρόταση. Για μας είναι πολύ σημαντική. Κύριε Πρέντεγκαστ, παρακαλώ, τα σχόλιά σας. Ξέρω ότι μεταξύ άλλων τα προκειμένα προσώπητα σας απασχολούν και σας ιδιαίτερα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή για αυτή την εξαντλητική παρουσίαση. Και εξής, κύριε Πρόεδρε, σε αυτά που είπατε και τη σημασία αυτής της πρότασης. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση, τη μάλλον την επιλογή εργαλείου που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε σχέση με την οδηγία του 99, ο κατακαιρματισμός των προτύπων ε, και θέματα δικαιοδοσία δείχνουν την ανάγκη για μία νέα ρύθμιση. Υπήρχαν κενά, σαφή αισθητά κενά. Και μάλιστα είχαμε μια τεχνική συνάντηση εδώ στο Βρυξέλλες, όπου παρατηρήσαμε μεγάλο ενδιαφέρον ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αν χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής αυτοποίησης, θα κερδίσουν πραγματικά τεράστιο χρόνο στη σύναψη συμβάσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, να εξαλειφθεί στο μέτρο του δυνατού η απάτη και από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη η τεχνική περιπλοκότητα του συστήματος θα δοθεί διαφορετικά από τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης με τα θέματα πληροφορικής ε, που έχουν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην καταλήξουμε σε λύσεις που να είναι πραγματικά πολύ δύσκολες για μικρούς ε, ενδιαφερόμενους εμπόρους και απλούς πολίτες. Η τυποποίηση, η λειτουργικότητα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο στόχο της ε, εσωτερικής αγοράς. Εγώ σήμερα είναι σαφές ότι τα πρότυπα στον τομέα έχουν απτυχθεί κατακρεματισμένα. Αυτό το είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο και πιστεύω ότι μια προσέγγιση με γνώμονα την ασφάλεια όπως χρησιμοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα με τις ε, τραπεζικές συναλλαγές ε, στο ίντερνετ δείχνουν πώς μπορούμε να επιτύχουμε και εδώ. Η πιστοποίηση των εγγράφων και τα ε, ηλεκτρονικά, ε, ηλεκτρονικές οροφές, ηλεκτρονικές κτλ. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη ρυθμιστικών μέτρων για να μπορούμε να, ενισχύσουμε τη χρήση αυτών των εργαλείων μέσω του διαδικτύου. Πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας της ε, επιγραμμικές συναλλαγές μέσω αυτο και ελπίζω να μπορέσουμε να μην έχουμε αρνητικό αντίκτυπο με υπερβολικές νομικές απαιτήσεις. Όπου δηλαδή ακόμη και σήμερα δεν θεωρείται αναγκαίο να έχουμε συστήματα λειτουργική αυτοποίησης σε τακτική βάση, δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε αυτά τα προσκόμματα στο μέλλον. Θα πρέπει η αρμόδιοι υποπτικοί ε, ε, φορείς σε εθνικό επίπεδο να έχουν το κατάλληλο δυναμικό και να παρακολουθούν τη συμμόρφωση ακολουθώντας τις ρυθμιστικές ε, διατάξεις της χώρας τους και με ό,τι αποφασίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, κατά 12 για άτομα αναπηρίες και την προσβασιμότητα. Μου φαίνεται αρκετά σαφές άρθρο και παρότι κατανοώ πρέπει να υπάρχει ευελιξία ταυτόχρονα Πιστεύω ότι το άρθρο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Έπειτα, η διάταξη για την συνεργασία με συμφωνίε που θα συζητώνται εξ ονόματο τη Ένωση, στηρώντα πλήρως την ασφάλεια και προστασία δεδομένων και την εποπτεία αυτών. Ω μέλο τη αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη σχέση με τη ΣΥΠΑ. Θέλω να επισημάνω ότι καθώ βάζουμε τα θεμέλια για οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητα με τη ΣΥΠΑ και να χρησιμοποιήσουμε τι εθνικέ στρατηγικέ για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματο με προκειμένου. Θέλουμε να θαρρύνουμε την Κομισιόν να είναι πάρα πολύ προσεκτική να δουλέψει και σε αυτό το μέτωπο παράλληλα με τις άλλες πτυχές της μελλοντικής συμφωνίας. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και για τα τεχνικά εμπόδια εγκαίρως για να μπορέσουμε να τα άρουμε. Μια τόσο καλή παρουσία. πιστεύω ότι έχουμε πολλές Ε, προσβλέπω συνεργασία με τον εισηγητή του Σκιώδη και με του συναδέλφους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο για τόσο σημαντική πρωτοβουλία, Πρόεδρε. Thank you um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εύστοχα αυτά που μα είπατε και ενδιαφέροντα. Πραγματικά θα είναι προκλητική όλη αυτή η δουλειά και με μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριο Κρότσμαν. Ο φίλος μου Μπουσόη με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω και το πράττω ευχαρίστω γιατί είμαι μάλιστα και σκιώδη συγητής στην αρμόδια επί της τη επιτροπή. Τέλο πάντων να μην μαλώσω με την κυρία Γκαλό, εδώ μπορεί να έχει άλλη άποψη για το ποιο πρέπει να είναι, ε, ποια πρέπει να είναι η αρμόδια επί τη επιτροπή. Πρόσφατα συζητήσαμε την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Εκτός από τα πρακτικά και ε, νομικά προβλήματα υπήρχε ένα πιο σημαντικό, την εμπιστοσύνη δηλαδή στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η προκείμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαφώς μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις και για τους καταναλωτές και για τους επιχειρηματίες. Αν και δημιουργήσαμε την απαραίτητη νομική βάση με την οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή, Αναγκαζόμαστε ωστόσο να διαπιστώσουμε ότι τα εθνικά συστήματα ποικίλουν, διαφέρουν πολύ σημαντικά και συχνά είναι ανεφάρμοστη η ηλεκτρονική υπογραφή. Συζητήσαμε και τις ηλεκτρονικές αναθέσεις, τις ηλεκτρονικές υποβολές προσφορών. Παρέτητο να μπορεί να πιστοποιείται ο υποβάλλον την προσφορά και αυτό ακόμη προκαλεί προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι, ότι προτείνοντας κανονισμό η Κομισιόν βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Για να υπάρξει ευρεία αποδοχή χρειάζεται και η δημιουργία της απαραίτητης εμπιστοσύνης. Εν προκειμένου το ερώτημα που θέτω εγώ είναι εάν τα συστήματα ταυτοποίησης δεν θα πρέπει να εξετάζονται από ανεξάρτητες αρχές. Η ευθύνη των χωρών μελών ενδεχομένως να εξισορροπεί κάποιες ελλείψεις, δεν αποκαθιστά όμω την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω πώς εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων στην πράξη. Πώς θα συμφωνήσουν ποιο θα χρειαστεί η ποια χώρα να προσαρμόσει το σύστημά τη και ποια όχι. Βέβαια για την διαλειτουργικότητα θα ρυθμιστούν τα πράγματα, ε, οι λεπτομέρειες δηλαδή, με εφαρμοστικές πράξεις της Κομισιόν, διότι ο κανονισμός περιλαμβάνει και πολλές εξουδοτήσεις για την Κομισιόν. Θα χρειαστεί να συζητηθεί εάν όλες αυτές οι εξουδοτήσεις είναι όντως απαραίτητες και εάν ορισμένα δεν θα πρέπει να τα ρυθμίσει ο ίδιος ο νομοθέτης. Ολοκληρώνοντας επανέρχομαι στην σημασία των υπηρεσιών αυτών για, πολι... για πολίτες και για επιχειρήσεις, για τη μείωση των διαμεθοριακών ε, στοιχείων κόστους των συναλλαγών. Πρέπει βεβαίως να είμαστε και προσεκτικοί. Να μην θίξουμε δηλαδή επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί ή αποφάσει αποφάσεις που, έχουν, που έχουν ληφθεί ήδη για μελλοντικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα το γερμανικό σύστημα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που βρίσκεται πραγματικά στο ε, πιο σύγχρονο επίπεδο της τεχνολογικής εξέλιξης. Άλλο θέμα είναι των ηλεκτρονικών σφραγίδων και πώς θα ενταχθούν στα εθνικά δικαιϊκά συστήματα. Άρα υπάρχει ακόμα ανάγκη συζητήσεως. Γι' αυτό χαίρομαι για την πρόταση της Κομισιόν και είμαι πεπισμένος ότι προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Μερικές παρατηρήσεις από μέρος μου. Πρώτον θεωρώ ότι είναι μια επίκαιρη και σωστή πρόταση. Πράγματι έχει βρει μια σωστή ισορροπία η Επιτροπή μεταξύ της ευθύνης σε εθνικό επίπεδο και τον, και τον κεντρικό συντονισμό. Ε, θα αποδεχθούν, ελπίζω, τα κρατημέλη αυτή τη λύση. Είχαμε πρόσφατα ζητήματα στον τομέα της ε, ψηφιακής ε, πολιτική κοινοποίηση, όπου τα κράτη-μέλη ε, ήταν μάλλον επιφυλακτικά στην ε, ύπαρξη κεντρικού συντονισμού σε τέτοια ζητήματα. Όμως είναι η μόνη πρακτική λύση. Γιατί υπάρχουν εξελίξει και στα κράτη-μέλη επιμέρου, όμω πλέον θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβή αναγνώριση. Και μάλιστα με επιτυχημένο τρόπο. Πρέπει να βρεθούν κάποια κίνητρα για να βάλουν πόρους σε αυτή την υπόθεση. Και αυτή είναι πάντα η δυσκολία. Και σε ό,τι αφορά την ε, εποπτεία, τα κράτη-μέλη δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ε, υπηρεσίες παρακολούθησης της εμπιστοσύνης, των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα στη σύνοψη. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει πρόταση το ε, εσωτερικό σύστημα πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς να είναι ένα ε, εργαλείο που να χρησιμοποιείται από τα γνωμοδοτικά αυτά όργανα, όπως χρησιμοποιείται σε άλλους τομείς. Γιατί στον κανονισμό IMI το έχουμε εντάξει αυτό. Ίσως κάνω λάθος βέβαια εδώ. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αυτές τις ε, πτυχές, να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα στα κρατη Και επίσης είδα ότι η Επιτροπή θέλει να υπάρξει κάποιος ε, δομημένος ε, πυρήνας συντονισμού ούτω ώστε αυτά τα εποπτικά όργανα να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ του. και να χειρίζονται καταστάσεις όπως η παραβιάση της ασφάλειας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 15 υπάρχουν ε, αναφορές ε, στις παραβιάσεις της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων πρέπει και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ζητήματα προστασία δεδομένων να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Όμω χαίρομαι που μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα την εξέταση αυτή τη πρόταση και είμαι σίγουρη ότι η κυρία Γκαλό θα κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει κάτι άλλο? Okay. Καλώς. Ε, υπάρχει κάτι άλλο από την εισηγήτρια, από την Επιτροπή. Επιτροπή. Ξέχασα να απαντήσω στην εισηγήτρια σε σχέση με την προστασία δεδομένων. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου αυτό το στοιχείο γιατί αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Η διάταξη λοιπόν λέει ότι όταν εγκατασταθεί αυτό το ε, πλαίσιο βεβαίω και θα είναι άμεσα εφαρμοστέο για τον κανονισμό. Πλέον όμως της αρχής του privacy by design. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουν, ε, θέλουν να παράσουμε με αυτές τις ε, υπηρεσίες εμπιστοσύνη. Ε, ιδίως ό,τι αφορά την ελοχιστοποίηση των δεδομένων, που είναι σημαντική η δικλίδα ασφαλείας. Τελευταίο σημείο αφορά τη διεθνή διάσταση Βεβαίω, ε, η ανάπτυξη τέτοιων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, είτε της κυβέρνησης είτε των ε, δημοσίων αρχών. άλλες ε, χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν κάποιον ιδιωτικό πάροχο τέτοιων υπηρεσιών που να θεωρείται ότι παρέχει επαρκείς ε, υπηρεσίες προς τον πολίτη. Έτσι μπαίνει το στοιχείο της υποχρεωτικής εποπτείας και έτσι αυτό δεν είναι εκτός ε, του πεδίου του κανονισμού κατά τη γνώμη μας. Γι' αυτό και έχουμε διατυπωθεί με αυτόν τον τρόπο το προκειμένο κεφάλαιο. Είναι ευθύνη των κρατών μελών, είναι πλήρης, πλήρως απόφαση δική τους. Βεβαίως διατηρούν την ε, διατήρηση της ε, συμβολής τους και της δέσμευσή τους είναι σημαντική. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο νομικό υπόβαθρο από τον κανονισμό ως προς την αξιολόγηση. Και εξετάζουμε διάφορα άλλα ενδιαφέροντα ε, πρότυπα για, για το πώς μπορούν αυτά τα πρότυπα να συνάδουν και με τα ε, επιμέρους ε, συστήματα ανακράτος μέλος. Αυτά τα στοιχεία ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστώ. would you like to just conclude... Κυρία Γκαλό, θα θέλατε να κάνετε κάποιες καταληπτικές παρατηρήσεις και να επιβεβαιώσετε και το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίω, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτον την Επιτροπή για τις εξηγήσεις της και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους και δεύτερον να προσδιορίσω ότι η προθεσμία καταβολής κατάθεσης ε, τροπολογιών είναι η 15η Μαΐου. Ευχαριστώ. Um, Στις 25 Απραλίου θα εξετάσουμε την έκθεσή σας. Πρέπει να τη στείλετε λοιπόν για μετάφραση μέχρι τις 4 Απριλίου. Έχετε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά σα. Ξέρω ότι θα τον αξιοποιήσετε σωστά. Τελική ψηφοφορία στις 9 Ιουλίου και η Επιτροπή Βιομηχανίας θα την ψηφίσει μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφου ε, από την Επιτροπή. Ε, οι διαφάνειες υπάρχουν και σε έντυπη μορφή, ε, αλλά θα τις βάλουμε και στο διαδικτύο. Ωραία, ας πέρασουμε στο τελευταίο σημείο της μέσας διάταξης για σήμερα. Σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. ευεργέτημα παινία σε διασυνοριακές πολιτικές και εμπορικές διαφορές. Βεβαίως αφορά τη δραστηριότητα ε, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, ιδίως ε, σε ό,τι αφορά τους πολίτες και, τους, ε, και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Ο Χάνς Πίτερ Μάγιαρ είναι εισηγητής. Η κυρία Πέρες είναι σκιώδης. Ξέρω ότι θα πάρει το λόγο λοιπόν. Και έχω και κάποιες σημειώσεις του κυρίου Φόξ. Από πλευράς Επιτροπής... Έχουμε την κυρία Σασταμόινεν, αν το προφέρω σωστά. Ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή? Ζεγόμου καριά το ονομάζομαι και αντικαθιστώ την ε, Διευθυντρία. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο στη συνέχεια. Κύριε Μάιερ, είστε έτοιμος. Μπορείτε να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας. Κυρία Πέρες, θα σχολιάσετε στη συνέχεια και εγώ θα προσθέσω κάποια στοιχεία εκ μέρους του κυρίου Φόξ. Και μετά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ. Sorry, I didn't notice. You're not on my list. Are you, are you the official shadow or the acting shadow? Hmm? You're the substantive shadow, are you? Officiel, yeah. far as you can Κύριε Ροσφόρ, είστε επίσημος ο Εσκιώδης ή ανεπίσημος. Καλά, θα μιλήσετε κι εσείς. Okay, ο κύριος Μάιερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση της Κομισιόν της 23ης Φεβρουαρίου πέρσι αναλύει την εφαρμογή της χρήσεως για την ενίσχυση για την αντιμετώπιση δικαστικών εξόδων που ισχύει από το 2004, δηλαδή 10 χρόνια περίπου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σχετικά λίγοι πολίτες και λίγοι ε, δικηγόροι άλλα σχετικά νομικά επαγγέλματα έχουν ποιήσει χρήση της δυνατότητας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό κυρίως για τους δεύτερους. διότι αυτό είναι παράδειγμα και για πολλούς άλλους τομείς της ε, πολιτικής δικονομίας. Η Κομισιόν η ίδια μιλεί εδώ και καλά λέει ότι χρειάζεται να γίνουν μικρές τροποποιήσεις στο σύστημα, αλλά η διαδικασία αυτή ισχύει από την 1η Πρώτου 2009 και έχει γίνει μελέτη μέχρι το 2010 και γι' αυτό δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο μέσα σε δύο χρόνια δεν μπόρεσαν δίθεν να υπάρξουν αποτελέσματα. Ένα σημαντικό ε, θέμα πρέπει να είναι κιόλας ότι η Κομισιόν παρακολουθεί, εποπτεύει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Η έκθεση της Κομισιόν διαπιστώνει σε τρία σημεία ότι η εφαρμογή σε ορισμένες χώρες μέλη τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς, δεν έχει επιτευχθεί. Και αυτό αφορά πρώτον τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των δικαστικών δαπανών, τα σχετικά έγγραφα και την κάλυψη των σχετικών εξόδων ταξιδιού. Είναι σημαντικά θέματα αυτά. Η σωστή λοιπόν εφαρμογή ε, μεταφορά στα εθνικά δίκαια έχει σημαντικό ρόλο να παίξει γιατί πρέπει να μπορεί να βασίζεται ο Ευρωπαίος πολίτης μέσα στα πλαίσια της μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς στις ρυθμίσεις αυτές και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα, μέτρα να γίνουν πραγματικές εκστρατείες διαφώτισης και να υπάρξει και ε, ένα data pool σε όλη την Ευρώπη, μια συγκέντρωση δηλαδή δεδομένων. Και εγώ αναμένω κυρίως την συνδρομή των νομικών επαγγελμάτων που διαθέτουν και τις απαραίτητες νομικές γνώσεις και να καταχωριστούν και στις σχετικές ε, γλώσσες τους. Έχουμε πολλές ε, δικονομικές διατάξεις. Έχουμε ε, επεξεργαζόμεθα μια κοινή ερμηνεία συμβάσεων. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής έχουμε εκτελεστικές διατάξεις, διατάξεις για επίδοση εγγράφων, έχουμε για καταδημολίες διαδικασίες το small claims, τη διαδικασία small claims των μικρών δηλαδή διαφορών, έχουμε για όλα αυτά και την χορήγηση του ευεργετήματος παινίας. Από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί κάποτε συμμετέσχουν σε μια διαδικασία small claim, δεν είναι γνωστά τα πράγματα αυτά ούτε καν στα δικαστήρια παρόλο που εδώ και πολλά χρόνια είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν τα σχετικά έγγραφα. Σε κάθε δικαστήριο πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο τον οποίο να μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες και να τους βοηθεί στην συμπλήρωση των εγγράφων. Βεβαίως και πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες και για ε, το ενδεχόμενο να λάβουν ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δικαστικών δαπανών. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες το Electronic Trust Service, δηλαδή η ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης, είναι σημαντική για την απλούστευση. Σε όλες τι διαδικασίες προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε. στι διαδικασίε των ε, μικρών διαφορών επήλθαν πολλές απλουστεύσεις και απέναντι στην γερμανική ε, πολιτική δικονομία. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται έγγραφα, χρειάζεται ανταλλαγές πληροφοριών και διαμεθοριακά. Σε τέτοιες διαδικασίες λοιπόν είναι απαραίτητο και σε αυτές να υπάρξει κάποια αξιόπιστη ηλεκτρονική διαδικασία για τη μείωση των ε, δαπανών, ε, των εξόδων δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Πέρασε για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμμερίζομαι πολλά από όσα είπε ο κύριος Μάγερ αναμφίβολα στο τομέα δικαιοσύνης ε, μένουν πάρα πολλά να κάνουμε, ιδιαίτερα στο το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη που είναι ακρογωνιαίος λήθος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας και με βάση όσα προβλέπει το άρθρο 47 του Χάρτη Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εγγυάται από το δικαίωμα και στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών δεν μπορούμε να επιτρέπουμε το κόστος ε, που απορρέει από τη συνεργό χαρακτήρα της διαφοράς δεν επιτρέπουν στον πολίτη να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Μόνο ο πολίτη θα μπορέσει να εμπιστευτεί πλήρως στην ιστορική αγορά που είναι ακρογωνίως λήθος του Ευρωπαϊκού Κοδήματος η οδηγία του 2003 με τον ορισμό ελάχιστων κοινών κανόνων για, την, για το ευεργέτημα παινίας σε την περίπτωση βιοσυνεριακών διαφόρων ήταν το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς θα μπορούσαν να ε, ε, προσφύγουν σαν δίκα μέσα σε όλη ε, στη δικαιοσύνη πάντοτε Πάντοτε όμω μπορεί να βελτιωθεί ε, η νομοθεσία. Συμφωνώ με τον κύριο Μάγερ ότι είναι λυπηρό το γεγονό ότι δεν είναι γνωστό ότι μπορεί κανείς να απολαύσει τη δικαιοσύνη δωρεάν σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού ε, κώδικα. Το τελευταίο ευρωγραμματρό έλεγε αυτό τον ε, μήνα μόλις το 1 τρίτο των πολιτών είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα που έχουν καθώς έχουν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα την επικοινωνία και την ενημέρωση και να βελτιώσουμε, να χρησιμοποιήσουμε μάλλον αυτό το εργαλείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές και για τους νομικούς, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στα οικονομικά κριτήρια για την παραχώρηση του ευεργετήματος παινίας. Όπως λέει το άρθρο 1 της Οδηγής του 2003, ε, υπάρχει εγγύηση για ε, δωρεάν δικαιοσύνη για άτομα που εν μέρει πλήρως δεν μπορούν να καταβάλουν ε, το κόστος της δίκης. Όμως το άρθρο 5 αυτή της οδηγία δεν διευκρινίζει ε, περισσότερα πράγματα, οπότε μπορεί να οδηγήσει σε κάποια σύγχυση σχετικά με το ποιο έχει δικαίωμα στο ευεργέτημα παινίας. Και άρα μπορεί τελικά να υπάρξει περιορισμό και να φυγεί ουσιαστικά και η ουσία αυτού του δικαιώματος ε, το οποίο το έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ακουστεί υπόθεση του σε ένα δικαστήριο. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση θα κάνω κάποιες τροπολογίες ε, στην ε, κτλ. τα λοιπά. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ ο κύριος Ροσφόρ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την λήψη της οδηγίας μας βοηθά να αποκτήσουμε ένα, μια καλή εικόνα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας. Βεβαίω να πούμε ότι έχει μεταφερθεί σωστά στην, ε, ε, στις εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχει Υπάρχουν βεβαίω κάποιε διαφοροποιήσει, αλλά υπάρχει και το πρώτο σημείο τη έκθεση του κυρίου Μαγέρα και το οποίο παρατηρούμε με μεγάλη λύπη και ανησυχία. Πρόκειται για έναν περίπλοκο μηχανισμό. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν αυτό το δικαίωμα, αλλά δυστυχώ είναι περίπλοκο. Θεωρώ ότι είναι καλό το σχέδιο γνωμοδότηση. Έχει συμπεριλάβει ενδιαφέρουσε προτάσει. Ε, τη στηρίζω, ιδίω ό,τι αφορά το, ε, αυτή τη δεξαμονή, δεξαμενή ε, νομικών που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν και προβλήματα πρακτικού προσδιορισμού αυτών των επαγγελμάτων. Θεωρώ όμω ότι αυτή η ομάδα νομικών συμβούλων ίσως θα πρέπει να λάβει μια κατάρτιση για κάποια ζητήματα που είναι αρκετά εξειδικευμένα. Ο εισηγητή προτείνει να υπάρχει μία αρχή ανακρατο μέλο, Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μου. Είναι μία τέτοια αρχή που τα αναλαμβάνει τέτοια ζητήματα. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε. Γιατί αν πάνω από όλα πρέπει να έχουμε και δύο αρχές σε κάθε κράτος μέλος, είναι τόσο περίπλοκο το σύστημα που θεωρώ πραγματικά απαραίτητο της απλούστευσης ύπαρξη δηλαδή μία και μόνο αρχής. Και αυτό όχι μόνο για τους ε, πολίτες, αλλά για όσους συμμετέχουν και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Για να ξέρουν και τι πρέπει να περιμένει, τι περιμένει ο κόσμος από εκείνους. Σε ό,τι αφορά την ε, προσβασιμότητα σωστές οι παρατηρήσεις σας. Βρήκαμε βέβαια κάποιες πληροφορίες και στην πύλη e-justice, όμως πάντα μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Και εδώ, κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης ανταλλαγής απόψεων, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα στον εισηγητή. Ε, παραπέμπει στην παράγραφο 7 αυτό που απορρέει από την αξιολόγηση τη επιτροπή, δηλαδή ότι πρέπει να λαμβάνουμε τα υπόψη το διαφορετικό κόστος ζωής στα κράτη-μέλη. Να γνωρίζουμε δηλαδή το κατόφλι που επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα τέτοιο επίδομα. Αυτό συμβαίνει ήδη, δηλαδή πρέπει έτσι κι αλλιώς να το κάνουμε, αλλά πώ το κάνουμε, ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια. Και από την άλλη ξέρουμε ότι ακόμα κι αν έχουμε τέτοια απριόρια αντικειμενικά κριτήρια, πρέπει ο ετών να ε, παράσχει και εγγραφά που αποδεικνύουν την οικονομική του ε, κατάσταση και όταν εμπλέκεται και ένα τρίτο κράτος μέλος δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο και κατά πόσο είναι εύκολο να επαληθεύεται και η εγκυρότητα αυτών των εγγράφων. Ίσως εδώ πέρα θα πρέπει να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Στην παράγραφο 8... Βεβαίω και πρέπει τα κράτη-μέλη να καταβάλουν περισσότερε προσπάθειε. Δεν κατανοώ γιατί ο κ. Μάιερ λέει αντίθετα από την Επιτροπή, γιατί υπάρχει αυτή η επίκριση εδώ. Ίσως ε, δεν έχω παρακολουθήσει καλά την ε, κατάσταση. Και τέλος, στην παράγραφο 10, ο κύριος Μάγερ μας λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί η αναρμόνιση των, ε, της νομοθεσίας των κρατών μελών με σκοπό να αποφευθούν περαιτέρω νομικά κενά. Πρέπει δηλαδή να πάμε προς την εναρμόνιση που είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να καταλάβω ως θέση του εισηγητή. Ότι μέχρι εκεί φτάνει δηλαδή αυτή η διατύπωση. Προφανώς ε, πρόκειται για διευκρινιστικά ερωτήματα, γιατί η ομάδα μου στηρίζει πλήρως το σχέδιο γνωμοδότησης και βεβαίω θέλουμε να συνεργαστούμε με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και να βοηθήσουμε για να συνδράμουμε την Επιτροπή Γιούρη στο έργο της. Ευχαριστώ. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Το ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα για το κύριο Μάγερ έχει αναλάβει αυτό το φάκελο δεδομένου της εμπειρίας του και εγώ δεν γνώριζα πολλά πράγματα μέχρι οπότε είδα αυτή την έκθεση ότι υπήρχε δυνατότητα ευεργετήματο παινία για α, αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Την έκθεση της Κομισιόν δεν την είδα, δεν την βρήκα. Δεν ξέρω δηλαδή ποιες θα είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων χρησιμοποιείται αυτό το ευεργέτημα παινίας. Εμείς που θέλουμε να λειτουργεί ομαλά η ενιαία αγορά και θέλουμε να ε, ασκούν τα δικαιώματα τους οι πολίτες σε μας απασχόλει. Και ε, έχουμε υπάρξει αρκετά ενεργοί να πείσουμε την Κομισιόν, τώρα το έκανε, να δημοσιεύσει έναν χάρτη για τα δικαιώματα του καταναλωτή στην ενιαία αγορά. Και μπορεί το κεντρικό βάρος να είναι η εσωτερική αγορά. Καλό θα ήταν να γίνει μια πιο ερετημνία στο δικό μας ε, έργο, δηλαδή ότι εστιάζουμε στον πολίτη, καταναλωτή. Μπορεί να σχολιάσει και η Επιτροπή αν το επιθυμεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι που εμείς ως Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς πρέπει να το δούμε ως προστιθέμενη αξία σε αυτήν την πρόταση. Το πρώτο μου σχόλιο ήταν αυτό. Και έπειτα να πω ότι γενικώ πώς. Επειδή έχουμε να κάνουμε μία έκθεση για το πώς έχουν τα πράγματα, ξέρετε, η Κομισιόν λέει μέσα που είναι σαφώς τα πράγματα πάνε καλά, μεν, αλλά από την άλλη τρέπεται να πει ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Όμως τελικά το επίπεδο δραστηριότητα είναι τόσο χαμηλό, οπότε δύσκολα μπορεί κανεί να έχει μια κατά πόσο τα πράγματα δεν είναι αποτελεσματικά ή δεν υπάρχουν δραστηριότητε γιατί οι πολίτε δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του ή γιατί φοβούνται τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε. ή για το πόσο δύσκολο είναι να βρει ένα δικηγόρο να κάνει καλά τη δουλειά του και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να τον πληρώσει δεν νομίζω ότι μας προσδορίζει καλά αυτό το έγγραφο προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι άλλο που παρατήρησα στις παρατηρήσεις της Επιτροπής η Επιτροπή κάνει κάποιες σκέψεις, μεν, αλλά δεν μιλάει για κάποιο σχέδιο δράση συγκεκριμένα. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι η δική μας η δουλειά θα έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Βλέπω πάντως μια πρόταση τώρα, η οδηγία αυτή να αλλάξει ουσιοδός ή να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ενεργητικά. Αυτές είναι κάποιες ε, σκέψεις του κυρίου Φόξ, που, ο οποίος μάλλον ως εξαιρετικός δικηγόρος θα μπορούσε να τα πει πολύ καλύτερα παρά τον τρόπο που τα λέω εγώ, ο οποίος δεν είμαι επαγίων. Υπάρχουν άλλα σχόλια πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή να τοποθετηθεί. Όχι. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτήν τόσο περιστατωμένη γνωμοδότηση. Μπορούμε να υιοθετήσουμε τις περισσότερες από τις προτάσεις του εισηγητή, γιατί και εμείς έχουμε τον ίδιο στόχο με εσάς, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Συμφωνώ, η έκθεση της Κομισιόν μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιητική. Και όπως είπατε, πρόεδρε, λείπουν κάποια στοιχεία σχετικά με την φύση των διαφορών για την οποία μπορεί να υπάρξει ευεργέτημα παινίας. Έχουμε δουλέψει και με αναδόχους και με κρατημέλη και δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία συγκεκριμένα για να μπορούμε να εντοπίσουμε κατά πόσο μία διαφορά είναι καθαρά εγχώρια, εσωτερική ή έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Πρακτικά όμως θα μπορούσε να είναι δυνατό ο πολίτης και ο συνήγορός του να απευθύνονται άμεσα στο δικαστήριο, την έδρα του το δικαστήριο, όπως έκανε πριν την εφαρμογή ε, αυτής της οδηγίας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολύ ικανοποιητικό γιατί υπάρχει το κόστος μετάφρασης, ε, υπάρχει το κόστος του συνηγόρου. Στόχος της πρότασης είναι να ε, εξαλειφθούν αυτές οι δαπάνες. Γιατί εν μέρη αυτές οι δαπάνες τις απορροφούν οι αρχές διαβίβασης, άλλο μέρος του κόστους η αρμόδια αρχή που ε, δίνει το ευεργέτημα παινίας, όπως και η μετάφραση μπορεί να γίνει από την αρμόδια διαβιβάζουσα αρχή. Αυτό λοιπόν το σύστημα που προτείνει η οδηγία, αν εφαρμοστεί συστηματικά, θα διευκολύνει σημαντικά ε, την δυνατότητα πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα άλλα κράτη-μέλη και τους πολίτες. Υπάρχει όμως θέμα ενημέρωσης. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα και μεταξύ των δικηγόρων. Δεν έχουν ιδέα για αυτή τη διαδικασία. Και είναι κρίμα γιατί οι λίγες προθεσμίες είναι υπέρ του πελάτη. Γιατί η διαβιβάζουσα αρχή έχει μέσα 15 μέρες διαθέσεις να διαβιβάσει ε, τα στοιχεία στην άλλη αρχή. Και τα δικαιώματα που απορρέπουν οδηγία. Κάθε δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα να χορηγήσει, να εγκρίνει την, το μου παινίας. Και έπειτα για το χρονοδιάγραμμα, ε, να πω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κινήσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δύο χρόνια είπατε δεν κάναμε τίποτα. Δεν είναι αλήθεια. Είχαμε μία συνάντηση με τους επιρρογνώμους των κρατών μελών. Για να τους ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της έκθεσης. Τα κράτη-μέλη δεν έδειξαν επιθυμία να αναθεωρήσουν οδηγία, αλλά ε, να συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή της. Τώρα, για κάποιες επιμέρους προτάσεις που περιλαμβάνεται στο σχέδιο γνωμοδότησή σας. Θα πω ότι εμείς δεν έχουμε καμία εξουσία να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, να ορίσουν μια ενιαία αρχή γιατί σε κάποια ομοσπονδιακά κράτη πρέπει να ορίζονται διαφορετικές αρχές όπως είναι στην Ισπανία, στη Γερμανία. Αυτό ε, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, είναι εθνική αρμοδιότητα ο ορισμός της αρχής. Και εξαρτάται από το εθνικό σύστημα της κάθε χώρας τον τρόπο τον οποίο ορίζονται τα του ευεργήματος περνίας. Συμφωνώ παντός μαζί σας κύριε Σεγητά. Θα μπορούσαμε κάποια στοιχεία από το website Atlas να τα συμπεριλάβουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, στο σχετικό πόρταλ. Ε, σε σχέση με τα έντυπα, συγκεκριμένα και τη διαθεσιμότητά του στο διαδίκτυο, ναι, υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Εγώ έκανα μια προσπάθεια να κάνω μια αίτηση για ευεργέτη με παινία στα γαλλικά. Στο έντυπο έβαλα το όνομά μου, πάτησα το κουμπί να μεταφραστεί στα αγγλικά, έγινε. Το σύστημα μου επέτρεψε είτε να κάνω αποθήκευση σε PDF ή να στείλω άμεσα σε email, με email προς το Ενωμένο Βασίλειο, π.χ ή στην Ιρλανδική Αρμόδια Αρχή. Οπότε μπορεί κάποιες χώρες να έχουν κάποια προβλήματα, μπορεί κάποιοι υπολογιστές να δημιουργούν πρόβλημα. Είναι τεχνικό το ζήτημα που μπορείτε να μας το κοινοποιήσετε για να δούμε τι είδους τεχνική λύση μπορούμε να δώσουμε. Είναι καλή αυτή η οδηγία, θεωρούμε, και ήταν ένα από τα πρώτα εργαλεία που εφαρμόστηκαν πρακτικά στο κεκτημένο του αστικού και εμπορικού δικαίου. Και ήδη υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών τέτοιων διαδικασιών και πάντοτε προκύπτει βεβαίω το ίδιο πρόβλημα, κατά πόσον στέφονται με επιτυχία ή όχι, γιατί έχουμε πολλές φορές 28 διαφορετικά δικαστικά καθεστώτα που έρχονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Θα πρέπει, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα επαρκώς ελκυστικό για τον ετούντα, ώστε να μπορεί να προσφύγει και σίγουρα να μην είναι μια διαδικασία που θα του επιφέρει ε, δυσανάλογο κόστος. Θα προσπαθήσουμε πάντω να ε, καλύψουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ελλείμματα που, όρισε, που εντόπισε και ο εισηγητή. Πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίε που μα δώσατε, λέει ο Πρόεδρο, Και σίγουρα θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη και ο εισηγητή. Κύριε εισηγητά, θέλετε να συνοψίσετε και να μα πείτε και το χρονοδιάγραμμα. Ähm, Ευχαριστώ. Σύντομη σύνοψη. Ευχαριστώ την Κομισιόν που απαντά στα επιχειρήματά μας. Ευχαριστώ και τους συνεισηγητές μου. Στην ουσία συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα λογικό και πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά πολύ λίγο γνωστό και επομένως χρησιμοποιείται και λίγο. Αυτό που θα βοηθήσει ωστόσο μόνο είναι να υπάρχει μια ενημερωτική εκστρατεία Εκεί βέβαια πρέπει να βάλει και το χέρι στην τσέπη η Κομισιόν και να αναγκάσει και όλα τις χώρες, τις χώρες μέλη και αυτές να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Διότι υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες, τις οποίες έχουμε ήδη δημιουργήσει, που ωστόσο δεν είναι γνωστές. Αν δεν γνωρίζω ότι μπορώ στην διαδικασία μικροδιαφορών να υποβάλω αγωγές και διαμεθοριακά μέχρι 2.000 ευρώ, δεν θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω και αυτή τη διαδικασία που σαφώς κοστίζει λιγότερο από μια συνήθη διαδικασία. Και στην πράξη τι γίνεται εάν έχω μια διαμεθοριακή διαφορά. Δεν γνωρίζω τα πράγματα. Πηγαίνω στον δικηγόρο και θα μου πει ίσως ο Γερμανός δικηγόρος «Α, πω, πω, τώρα Ισπανία, Ελλάδα, πρέπει να πας να βρεις δικηγόρο επιτόπου». Τότε αυτός θα σας πει θα έρθει σε επαφή με κάποιο δικηγόρο λοιπόν επιτόπου, θα σα πει ευχαρίστω να αναλάβω την υπόθεσή σα, αλλά θα μου προκαταβάλλετε 2.000 ευρώ. Να λοιπόν, δεν μα βοηθήσει τίποτα αυτό. Η ενημέρωση είναι το σημαντικότερο όλων. Υπάρχουν βέβαια και άλλε σημαντικέ λεπτομέρειε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ανάλυση. Δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίε για το τι άλλο θα πρέπει να συμπληρωθεί. Χαίρομαι πάντω που η Κομισιόν έχει εντοπίσει πολλά, πολλές από τις ε, πτυχές όπως και οι συνεισηγητές μου. Δεν έχω λοιπόν καμία αντίρρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει και τουλάχιστον σε τρία μέρη ότι δεν έχουν πλήρως ε, μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια οι απαραίτητες διατάξεις. Εν πάση περιπτώσει μην εισμονείτε έχουν περάσει 10 χρόνια. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα έπρεπε να έχει γίνει γνωστή η διαδικασία αυτή και να λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να επιμείνουμε. Δεν επιτρέπεται να το δεχθούμε από την ε, εισαγωγή της διαδικασίας μικροδιαφορών, small claims, έχει περάσει πάλι μια τετραετία. Και αυτή δεν είναι γνωστή. Δημιουργούμε δικονομικές δυνατότητες για ε, να διευκολύνουμε τους πολίτες, πρέπει και να γίνουν γνωστές. Είναι βέβαια σαφές να έχουμε υπόψη μας και τα σχετικά δεδομένα. Για μας στη Γερμανία αρμόδια είναι τα ειρηνοδικεία. Πόσες τέτοιες υποθέσεις καλούνται να εκδικάσουν ε, τα δικαστήρια αυτά είτε εντός της επικρατείας είτε και διαμεθοριακά. Είναι πολύ δύσκολο. Το ίδιο και ακόμη περισσότερο για το ευεργέτημα παινίας που ούτως ή άλλως είναι διαδικασία δευτερεύουσα ως προς την κύρια διαδικασία. Τα έγγραφα ή τα έντυπα και εδώ είναι δυνατόν να υπάρξει ε, σημαντική βελτίωση. Εάν, για παράδειγμα, συμπληρώσω το έντυπο ως PDF στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχω όλα τα έντυπα αναχείρας, γιατί αλλιώ δεν μπορώ να το συμπληρώσω το ηλεκτρονικό έντυπο. Και αν λείπει έστω και μία πληροφορία, τότε καταραίει το όλον. Άρα πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή. Πολύ πιο λογικό λοιπόν θα ήταν αν μπορούσε να γίνει με τη μορφή ενός εγγράφου Word, πάλι, μιλώ πάντα για τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής, ώστε να μπορέσει να αποθηκευτεί και να επανέλθω να το συμπληρώσω όταν θα έχω στη διάθεσή μου όλα τα σχετικά έγγραφα. Νομίζω ότι τον Απρίλιο πρέπει να επανέλθουμε για να υποβάλουμε και νέες σκέψεις και προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα το απόγευμα. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 4 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, από τις 3 έως τις 6.30. Η Επίτροπος Ρέντινγκ θα είναι μαζί μας. Κύριε Μάγερ, σίγουρα θα είστε εδώ για να την ανακρίνετε εντό εισαγωγικών και για, αυτή την υπόθεση και για άλλε. Θα αναφερθούμε σε συζητήματα που αφορούν ε, την αγορά ενέργειας. Και μετά, κύρια συνάντηση θα είναι στις 20 και στις 21 Μαρτίου. Α, συγγνώμη, μάλλον ξέχασα το χρονοδιάγραμμά σας. Συγγνώμη που πανέρχομαι έχουμε πολύ σύντομη προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Μόνο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, το, σημείο σημειώνω αυτό. Σωστά. Και θα τις εξετάσουμε 21 Μαρτίου στη δεύτερη συνάντηση και θα ψηφίσουμε στις 11 Απριλίου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.